ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτους δικαίου και δημοκρατίας. Ξεκινάμε με το θέμα κατάσταση των ακτιβισμών των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Καμπότζη και το Λάος. Ξεκινάμε με την κυρία Σαρτζεντίνη μεταξύ των συντακτών του ψηφίσματος για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ εκ μέρους των Πρασίνων να αναφερθώ στο θέμα αυτό και στην παραγωγή ζάχαρη στην Καμπότζη και στο Λάος. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε γιατί υπάρχει αυτή η χειραγώγηση και γιατί υπάρχει τόσο κακή μεταχείριση των ε, κατοίκων εκεί. Γι' αυτό λοιπόν, εξού και το ψήφισμα αυτό, ελάχιστος μισθός στην κλωστεφαντουργία στην Καμπότζη είναι το 1 τέταρτο, οπότε θα έπρεπε να είναι ένας μισθό για να μπορούν να ζήσουν οι άντρες και οι γυναίκες εκεί. Πώς λοιπόν θα μπορέσουν να συντηρήσουν τι οικογένειε τους. Η εκμετάλλευση γίνεται μέσω βίέ και είναι καθημερινό φαινόμενο. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία που στηρίζει η γερμανική και η ολλανδική κυβέρνηση είναι προς την κατεύθυνση μισθών αξιοπρεπών και γι' αυτό και πιέζουμε για βιώσιμη παραγωγή, αξιοπρεπή παραγωγή που να μείβεται δηλαδή αξιοπρεπώς. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη διαφορά. Τώρα στα ζαχαρότεφλα. Εδώ βλέπουμε να αυξάνεται η παραγωγή στην Καμποτζή και στο Λάος κατά πολύ και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Όμως απαλατριώνονται τα κτήματα των κατοίκων πολλές φορές και αυτό είναι μία βία και χρησιμοποιούνται είτε γελμονάδες είτε για την κοκακόλα και αυτό θα έπρεπε να απαγορεύεται. Συνεπώς, Πρόεδρε, το καλό νέο είναι ότι η coca είπε ότι όχι, δεν θα συμμετέχω πια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κυρία Ντεκέζερ, για ένα λεπτό έχει το τον προηγούμενο Ιούλιο μετά από ε, εκλογές ε, οι οποίες ε, ήταν διάτρετες από απάτες ξεκίνησε μια ένα κύμα ταραχών στην Καμπότζη, οι οποίες, ε, ε, οι οποίες κατεστάλησαν με βίο τρόπο, κυρίως ε, οι τελευταίες, οι οποίες αφορούσαν τη διαμαρτυρία των εργαζόμενων στην κλωστοϊφαντουργία. Μεγάλες ευρωπαϊκές μάρκες έχουν υπεργολαβίες στις χώρες αυτές και είδαμε διαδηλώσεις με τις οποίες οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πύρ με πραγματικά πυρά. Ε, όπως είπε και η κυρία Σαργεντίνη, θα πρέπει εμείς σαν Ευρωπαίοι να έχουμε, να αναλάβουμε την ευθύνη του εμπορίου που κάνουμε ε, με τις ε, απάνθρωπες συνθήκες που ισχύουν στο, στην Καμπότζη και στο Λάος θα πρέπει να γίνουν συμφωνίες όπως αυτές ε, που ε, ξεκίνησαν και στο Μπαγκλαντές. Ε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε. καλούμε και την κυβέρνηση να ξεκινήσουν κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να ξαναβρεθεί η σταθερότητα στη χώρα. Και ζητούμε να γίνει διεθνής έρευνα όσον αφορά τις απάτες των τελευταίων εκλογών. Ευχαριστώ κυρία Σάκη, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών στην Καμπότζη. Οι εκλογέ έγιναν στο μέσο ατασταλιών και θα πρέπει να ερευνηθούν. Επίση, υπήρξε βία καταστολή των ε, ε, διαδηλώσεων με έξι νεκρού και πολλού τραυματισμένου. Ζητούμε από την κυβέρνηση να ελευθερώσει αυτού οι οποίοι έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και να διατηρήσει την ελευθερία του συνέρχεστα. Είναι απαραίτητο όχι μόνο να χαρακτηριθούν η υποχρέωση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά μπορεί η αντιπολίτευση να παίξει τον θεμητό τη ρόλο στην Καμπότζη. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια πολυμορφική πολιτική σκηνή για την ανάπτυξη τη χώρα αυτή. Ω Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα θέματα στο πλαίσιο συμφωνίες για γενικευμένες προτιμήσεις. Θα πρέπει να παραοτρύνουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν παραγωγή στην Καμπότση να δίνουν σωστές αμοιβέ στους εργαζομένους ώστε να μπορούν να επιβιώσουν. Και η κυβέρνηση Χανσέγκ θα πρέπει να σεβαστεί το δικό της το δικό του σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει. Για το λαός τώρα εξακολουθούμε να ανησυχούμε πάρα πολύ για την κατάσταση των ανθρωπινών δικαιωμάτων εκεί και παροτρύνουμε την κυβέρνηση να αναφέρει ποια είναι η, η κατάσταση του ακτιβιστή σώματο Ομπόνε, του ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι οδήγησαν στην εκούσια εξαφάνισή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κύριε για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο που εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάμε ψήφισμα σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο, τον Σόμπατ Σόμφων. Ο Σόμπατ απήχθη στις 15 Δεκεμβρίου του 2012 μπροστά από αστυνομικό τμήμα στην πρωτεύουσα του Λάος, το Βιετσίν. Κανείς δεν τον έχει δει από τότε. Γιατί το ξανασυζητάμε. Διότι πριν από την εξαφάνιση, εκείνος δούλευε ειρηνικά για να προωθήσει την προστασία του περιβάλλοντος και την εκπαίδευση στη χώρα του. Ήταν ένας από αυτούς που οργάνωσαν το φόρουμ που έλαβε χώρα στο Βιέντσιμ λίγο πριν από την εξαφάνισή του. Συζητάμε επίσης το θέμα αυτό γιατί ο Σόμπατ αποτελεί σύμβολο για πολλούς οι οποίοι δουλεύουν προκειμένου να βελτιώσουν την κατάσταση ζωής των κατοίκων του Λάος. Δυστυχώς όμως υπάρχει μεγάλη καταστολή. Οι αρχές του Λάος προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε την εξαφάνιση αυτή του Σόμπατ. Καθυστερούν, αρνούνται να αναλάβουν βήματα προκειμένου να λύσουν την υπόθεση αυτή. Το διαπίστωσα και προσωπικά όταν επισκέφτηκα το φθινόπωρο ίδιο στο Λάος. Σε ένα mail της προηγούμενης εβδομάδας, η πρεσβεία του Λάος στις Βρυξέλλες παραδέχτηκε ότι η πιο πρόσφατη αναφορά σχετικά με την υπόθεση είναι του Ιουνίου του 2013, δηλαδή πριν από πάνω από έξι μήνες. Αυτό είναι σκανδαλώδες. Το ψήφισμά μας λοιπόν ζητάει δράση, να αναλυφθεί δράση. Αποσαφηνίζουμε ότι δεν έχει λυθεί η υπόθεση αυτή, κάτι το οποίο εμποδίζει το Λάος να γίνει μέλος του Συμβουλίου σχετικά με τα θέματα αυτά στα Ηνωμένα Έθνη. Πιστεύω ότι πρέπει να στείλουμε την υποστήριξή μας στην οικογένειά του και σε όλους όσοι αγωνίζονται για τα δικαιώματα αυτά. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ευχαριστώ. Ακολουθεί για να κύριο Στάνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εξουσία στην Καμπότζη είναι 27 ετών και το Λάος έχει κομμουνιστική κυβέρνηση με τρεις ηγέτες τα τελευταία 7 χρόνια. Όλα αυτά οδηγούν σε μια κατάσταση εδραίωσης της ένδυας και όχι εξυπηρέτησης της ανάγκης των πολιτών οι ε, διαδηλώσει οι οποίε έγιναν στην Καμπότση έχουν οδηγήσει σε βία και καταστολή από την πλευρά τη κυβέρνηση και η κατάσταση αυτή φαίνεται να συνεχίζεται και το 2014. Είδαμε πέντε εργαζόμενου σε εργοστάσιο ένδυσης να σκοτωθούν από τι δυνάμει ασφαλεία τη κυβέρνησης και στο γειτονικό λαός που είναι κομμουνιστική δικτατορία. Η εξαφάνιση ενό ηγέτη τη κοινωνία των πολιτών και ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Σόμπατ και το γεγονός ότι οι αρχές του Λάους δεν θέλουν να διερευνήσουν αυτή την υπόθεση και να δεχτούν διεθνή συμφωνία, διεθνή βοήθεια για κάτι τέτοιο, αυτό μας κάνει να ανησυχούμε. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τονίσει περισσότερο την ερασιμότητα επί τη βάση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν δίνει βοήθεια αναπτυξιακή στις χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνοκ. Ο κύριος Λίζεκ για ένα μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ θετικό ότι βλέπουμε και πάλι την κατάσταση στην Καμπότζη και το Λάος. Γιατί η κατάσταση είναι απόλυτα απαράδεκτη σε όλους μας. Μετά από τις πρόσφατες εκλογές, οι οποίες δεν τηρούσαν τα διεθνή πρότυπα, ακολούθησαν μαζικές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες. και επίσης λόγω της, πολιτικ... λόγω της πολιτικής κατάστασης αλλά λόγω και της εξατλειωτικής κατάστασης των στα εργοστάσια ένδυσης. Υπήρξε φόνος ενός αριθμού διαδηλωτών και ακτιβιστών από την αστυνομία και τραυματισμός πολλών ατόμων. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν, πρέπει να τονίσουμε το πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα αυτά και να καλέσουμε την κυβέρνηση της Καμπότζης να βελτιώσει την κατάσταση, να έρθει σε επαφή με την αντιπολίτευση και να αποζημιώσει αυτούς που τραυματίστηκαν. Πρέπει να υπάρξει και παρακολούθηση από την ύπατη εκπρόσωπο της κατάστασης αυτής και να αναλάβει δράση και ο ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή για το Λάος, νομίζω. Και εκεί θα πρέπει να υπάρξει διευκρίνηση των συνδικών εξαφάνισης του κ. Σομπάτ Σομφών από την κυβέρνηση του Λάος. Ευχαριστώ κύριε Λίσε. Ακολουθεί η κυρία Εσαϊά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε έχουμε ε, την Καμπότζη και το Λάος και οι δύο χώρες ε, διανύουν ανησυχητικές περιόδους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, βλέπουμε επίσης και όλα τα προβλήματα τα οποία συνδέονται με εργασιακά ζητήματα. Στην Καμπότζη ας πούμε, Στην Καμπότζη έχουμε ε, τους συλληφθέντες μετά από τις διαδηλώσεις του μηνός Ιανουαρίου. Ήταν εργάτες οι οποίοι ζητούσαν απλώς αύξηση του μισθού του μισθού τους. Ε, οι δυνάμεις ε, ασφαλείας ε, καταχράστηκαν τις εξουσίες που έχουν με αποτέλεσμα δολοφονίες και τραυματισμούς. Στο ψήφισμά μας επίσης όσον αφορά το Λάος υπενθυμίζουμε ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε την υπόθεση του Σόμπα Θεσομπόουν ο οποίος ήταν ακτιβιστής ανθρωπίνων και λοιπόν δικαιωμάτων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσαφινιστούν τα πράγματα και να ξέρουμε πού είναι ο άνθρωπος αυτός. Η κυρία Σένσιν για ένα λεπτό ακολουθεί. Χωρίς, χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπουμε ε, στις χώρες αυτές ε, ανθρώπους που ζουν σε απόλυτη φτώχεια και μιζέρια, που ε, έχουν μισθό ένα δολάριο την ημέρα. Την 3η Ιανουαρίου σε ειρηνικές διαδηλώσεις εργαζομένων επενέβησαν οι δυνάμεις ασφαλείας, άνοιξαν πύρ και αφαίρεσαν τη ζωή πέντε ανθρώπων και τραυμάτισαν πολλούς περισσότερους. Θα πρέπει να το δούμε το ζήτημα αυτό, να χρησιμοποιήσουμε, να αναλύσουμε επίσης την χρήση των πυροβόλων ε, όπλων ε, και στην περίπτωση του Λάος ε, θα πρέπει να ζητήσουμε ο ακτιβιτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να απελευθερωθεί, να ξέρουμε την τύχη του και επίσης να υπάρξει και αποσαφήνιση των εκλογών του προηγούμενου έτος τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Το δικαίωμα στην ε, ιδιοκτησία γης επίσης ε, θα πρέπει να γίνεται σεβαστό. Διαφορετικά θα πρέπει να υπάρξουν ε, διαφοροποίησεις όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Καμπότζη και το ίδιο ισχύει και για τον Λάος. Σας ευχαριστώ. Θέλω να παρακαλέσω πάλι τους συναδέλφου να μην διαβάζουν τόσο γρήγορα κείμενα που οι διερμηνείς δεν μπορούν να τους προλάβουν. Εφόσον θέλετε να ακούσουν και οι άλλοι και να καταλάβουν αυτά τα οποία λέτε, θα είχε πιο πολύ νόημα να μιλάτε με χαμηλότερη ταχύτητα για να μπορέσει να υπάρξει πλήρης διερμηνία. Ο κύριος Μπένιον για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περίπου ένα χρόνο μίλησα για την κατάσταση στο Λάος και την ε, απαγωγή του κύριου Σαμπών στην Ολομέλεια αυτή, αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα έκτοτε. Εξακολουθεί να είναι άγνωστε οι συνθήκε τη απαγωγή. Και στην Καμπότση η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερα μετά από την καταστολή των δυνάμεων ασφαλεία κατά των εργαζομένων που έχουν κατέβει σε διαδηλώσει μετά τι κατά πάσα πιθανότητα ε, νοθευμένε εκλογέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει κατεπηγόντω να λάβει υπόψη την αξιολόγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την περιοχή, γιατί δεν μπορεί να δίνει προνόμια η Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρες οι οποίες εκδιώκουν ε, αγρότες από τα σπίτια τους χωρίς καμία αποζημίωση. Οι φιλελεύθεροι και οι δημοκράτες ζητούν να υπάρξει μια αίτηση δήλωσης από την πλευρά της Καμπότσης ότι δεν μάλλον από τις εταιρείες ευρωπαϊκές στην περιοχή να δηλώνω ότι δεν, η δραστηριότητα δεν οδήγησε στην εκδίωξη κανένας από το σπίτι του χωρίς αποζημίωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπένιον. Για ένα λεπτό. Ε, ο κύριος Μιγκάλσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Δεν ακούσαμε αρκετά ότι πριν από μερικούς μήνες είχαμε ξαναδεί και ξανεξετάσει την περίπτωση αυτή του κυρίου Σόμπατ ε, Σομφών. Αλλά ακριβώς αυτό περιμένουν και οι υπεύθυνοι. Εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε τις εκκλήσεις μας, να ζητάμε και να ξαναρωτάμε τι συμβαίνει, ώστε να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα του ανθρώπου αυτού. Αυτό λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε και στην περίπτωση τη Καμπότζη και του λαού, να επιμείνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί. Και πιστεύω ότι πρέπει να απαιτήσουμε όλες, να συνεχίσουν να κάνουν όλε τι προσπάθειε που είναι δυνατόν και εμείς να συνεχίσουμε τις δικές μας τις προσπάθειες, αλλά και όλες οι χώρες μέλη μεμονωμένα, αλλά και η κυρία Στονή είπα, Πρέπει να βοηθήσουμε τους υποστηρικτές, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές που έχουν ανάγκη και από ηλική και από ηθική βοήθεια. Ευχαριστώ. Μερσή κύριε Για 1,5 λεπτό κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι. Από ό,τι φαίνεται σε πολλές δημοκρατικές χώρες καλούμεθα να υποστηρίξουμε τα δημοκρατικά κινήματα. Πρέπει λοιπόν να εξηγούμε στους πολιτικούς επιτόπου ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο λόγος δηλαδή για τον οποίο του στηρίζουμε, είναι για να βοηθήσουν και αυτοί στην οικοδόμηση μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Οι παρεμβάσεις που γίνονται κατά των διαδηλωτών ή των εκπροσώπων στον κλάδο της κλωστιφαντουργίας αποτελεί μια αποτυχία των εκεί κυβερνήσεων που δεν δικαιολογείται με τίποτα. Ο εκφοβισμός του πληθυσμού, η χειραγώγηση των εκλογικών αποτελεσμάτων είναι πράγματα που δεν μπορούμε να ανοιχθούμε. Όπου και αν αυτά συμβαίνουν. Εμείς πρέπει να επηρεάζουμε και πολιτικά και οικονομικά και έτσι να προσπαθήσουμε να αλλάξει η κατάσταση και να προσφέρουμε καλύτερες προϋποθέσεις στους εργαζόμενους στην κλωστεφαντουργία εκεί. Είναι αναγκαίο η παραγωγή τους να πουλιέται στα μέρη μας. Νομίζω ότι μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τη διπλωματία μας και να επικοινωνήσουμε καλύτερα με τους πολιτικούς ηγέτες εκεί για να υπάρχουν λιγότερες συγκρούσεις. Κύριος Κλάς για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Το Λάος είναι μια σοσιαλιστική χώρα. Η Καμπότζα από την Human Rights Watch περιγράφεται σαν μια σαφής κομμουνιστική χώρα με αυταρχική κυβέρνηση η οποία λειτουργεί με επιφανειακή μονοδημοκρατία. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τον σοσιαλισμό εκεί, πώς ε, λειτουργεί, που τελικά υπονομεύει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποτέ στην ιστορία δεν κατέφεραν οι κομμουνιστές να κάνουν την ιδεολογία του να συνάδει με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι εργαζόμενοι τυχαίνουν εκμετάλλευση πολύ μεγαλύτερη στι κομμουνιστικέ χώρε. Και είναι αξιοπρόσεκτο αυτό για μια ιδεολογία η οποία στην ουσία θέλει να υποστηρίζει τους εργαζόμενους. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Κίνα, το βλέπουμε και στην Καμπότζη, το βλέπουμε στην κλωστιφαντουργία όπου είναι ματήρη πραγματικά η εκμετάλλευση. Άλλοι θανατώνονται, άλλοι τραυματίζονται και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες που βρίσκονται στις φυλακές. Δύο πράγματα λοιπόν πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε σαν πλατφόρμα την ΑΣΕΑΝ για να καταγγείλουμε τα γεγονότα αυτά και δεύτερον πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις στις χώρες αυτές. Να μην τους δίνουμε αναπτυξιακή βοήθεια όσο εξακολουθούν να υπάρχουν εκεί αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακολουθεί για ένα λεπτό η κυρία Κορχολά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα μέλη της ε, αντιπολίτευσης ήρθαν σε επαφή μαζί μας τον μήνα Σεπτέμβριο ε, και γνωρίζετε ότι δέχονται πάντοτε, και αυτό είναι σαφές, ε, πολλές απειλές. Τίποτα το δημοκρατικό δεν υπάρχει εδώ. Τα μέλη των συνδικάτων, τα μέλη της αντιπολίτευσης υφίστανται τρομερή πίεση. Ε, και επομένως ε, τι γίνεται με την ανεξαρτησία τους. Ε, στις χώρες που μας απασχολούν η αντιπολίτευση θεωρήθηκε υπεύθυνη για τις διαμαρτυρίες οι οποίες οργανώθηκαν ενώ δεν είχε καμία σχέση με αυτές. Πιστεύουμε ότι ε, ε, τα 23 μέλη των συνδικάτων που, που έχουν φυλακιστεί θα πρέπει να ελευθερωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα και μια έρευνα ε, ανεξάρτητη και διαφανής θα πρέπει να γίνει στην Καμπότζη από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κορχόλα. Θα δώσω το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Στίβενσον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ. Τι είναι συζήτηση για κατεπήγοντα ζητήματα. Αλλά η τραγική απαγωγή του κυρίου Σούμπαθ Σομχόουν ε, ξανασυζητήθηκε στην ε, Ολομέλεια. Ε, η καταστολή των εργαζόμενων στην εκλοστοϊφαντουργία στην Καμπότζη δεν είναι κάτι που πρέπει να αγνοήσουμε βέβαια αλλά ας δούμε λίγο ε, τα πράγματα λογικά. Ε, είχαμε ε, από την 1η Σεπτεμβρίου 7 απαχθέντες, εκ των οποίων 6 γυναίκες που ακόμα αγνοείται πλήρως η τύχη τους και δεν ξέρουμε τίποτα για αυτούς. Έχουμε την κατάσταση στη Συρία, έχουμε δολοφορίες και βομβιστικές απόπειρες στην Βηρητό, στην Βαγδάτη και δεν κάνουμε τίποτα και συζητάμε τούτα εδώ σαν κατεπήγοντα ζητήματα. Ας έχουμε λίγο την αίσθηση τη αναλογία, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Στίβενσον. Περνάμε στη διαδικασία HDI και δίνω το λόγο στον κύριο Κούκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να υποστηρίξω το έργο των ακτιβιστών στην Καμπότση και στο Λάος. Είναι απόλυτα απαραίτητο να μπορέσουν να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών. Πρέπει να τύχουν τις πλήρους προσοχής μας σε ό,τι αφορά την εργασία τους και, την... και θα πρέπει να προστατευτούν από οποιαδήποτε μορφή βίας εναντίον τους και θα πρέπει να είναι ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Υπήρξαν ταραχές στην Καμπότζη όπου σκοτώθηκαν άτομα. Οι εκλογές ήταν μεν καθαρές, αλλά θέλω να ζητήσω από τους πολιτικούς αρχηγούς να ερευνήσουν για κάποιες ατασταλίες που είναι κατά τη διάρκεια των ε, εκλογών αυτών. Και να πρέπει να υπάρξει διαλεύκανση αυτό το των γεγονότων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούκαν. Ο κύριος Ταραμπέλα. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, και εγώ λυπούμε που ανακατέψαμε λίγο τα πράγματα. Ε, η περίπτωση του λαούς και του Σομπάθου Σομφών οπωσδήποτε ε, είναι ε, πολύ σημαντικό. Αλλά εάν πρόκειται να πάρουμε την περιοχή σαν γεωγραφική, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι και για το Βιετνάμ. Η Καμπότζη όμω, αντιθέτω, πρέπει να μα ενδιαφέρει. Στι 3 Ιανουαρίου του 2014, εργαζόμενοι στην κλωστιφαντουργικό τομέα κατέβηκαν στο δρόμο ε, ζητώντα αύξηση μισθών. Οι δυνάμει ασφαλεία λοιπόν άνοιξαν ε, πυρ, ε, δολοφόνησαν πέντε ανθρώπου, τραυμάτισαν περισσότερου και οι άνθρωποι αυτοί ζητούσαν απλώ καλύτερε συνθήκε εργασία. Αυτό είναι απαράδεκτο γιατί η ελευθερία του εκδηλώνει ναι, και του του ελευθέρου συνεταιρίζεστε ε, είναι εγγεγραμμένη στο Σύνταγμα της ε, Καμπότζης ε, και επομένως πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που υπεραμείνονται των δικαιωμάτων των εργαζομένων να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν και θα πρέπει μέσω του ψηφίσματός μας να τους βοηθήσουμε κυρίως δε που δουλεύουν για πολυεθνικές εταιρείες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ταραμπέλα. Ευχαριστώ Κύριε Γιάχτερ Μακή για να κλείσει η συζήτηση. Arvoisa puhemies. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι εργαζόμενοι του εργαστηρίου ένδυσης που έχουν τύχει καταπάτηση των δικαιωμάτων τους σε πάρα πολλές χώρες. Και είναι χώρες από τις οποίες προμηθεύονται τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα. Κοιτάξτε τα ρούχα που φοράτε. Πολλά από αυτά ίσως έχουν φτιαχτεί στην Καμπότζη. Από την πλευρά της Κομισιόν ίσως έχει υπάρξει και κάποια σκέψη σε σχέση με αυτά τα προϊόντα. Πώς παράγονται, σε ποιες συνθήκες παράγονται που έρχονται από μακρινές χώρες αυτά τα προϊόντα. Είμαστε σίγουροι ότι τα προϊόντα αυτά είναι καταρχήν προϊόντα ποιότητος και δεύτερον τι έχει γίνει με τα δικαιώματα των ατόμων που έχουν παραγάγει αυτά τα προϊόντα σε ποιες συνθήκες έχουν εργαστεί αυτά τα άτομα. Γιατί έχουμε και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εργάζονται εκεί και οι οποίες πρέπει να ελέγχονται από την Ευρώπη. Δίνω τώρα το λόγο στον Επίτροπο κύριο Κάλλας. Mr. President, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η έγκριση κατεπήγοντα ψηφίσματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση στην Καμπότζη και το λαό μα απασχολεί σήμερα. Όσον αφορά την ε, Καμπότζη, ε, έγιναν εκλογέ τον Ιούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επέμεινε ώστε το δικαίωμα του συνδιαλέγεστε και του συναθρίζεστε και η αρχή της ελεύθερη επιλογής να ε, αναγνωριστούν. Ε, και επίσης ε, έκανε έκκληση η Ευρωπαϊκή Ένωση προς όλα τα κόμματα να συνεργαστούν και να βρουν μια λύση σε αυτό το πολιτικό αδιέξοδο. Όσον αφορά τα τελευταία συμβάντα της Δευτέρας και Τρίτης ε, Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει βαθύτατη, ε, βαθύτο προβληματισμό όσον αφορά κυρίως ε, την βία που έδειξε η δυνάμεις ασφαλείας και που κατέληξε σε αφαίρεση ανθρωπίνων ζώων. Επίσης όσον αφορά και την σύλληψη των ηγετών της αντιπολίτευσης Σαμ Ρέινση και Κέμ Σόκα έγινε μια ε, προσπάθεια να έρθουμε, ε, ε, μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ο Σαμ Μαρέινς έλεγε αμνηστή από τον εισαγγελέα της, του Βασιλείου 14 Ιουλίου και είχε την δυνατότητα να επιστρέψει στην Καμπότζη, παρόλα αυτά δεν είχε τη δυνατότητα να μας εντάξει στις εκλογές. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ξαναρχίσει ο πολύ ευάλωτος κοινωνικός διάλογος στην Καμπότζη. Μέσω της ε, μόνιμης αντιπροσωπείας της η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι, προσπαθεί να παίξει ρόλο στην ε, Καμπότζη. Είναι ένας από τους κύριους πρωταγωνιστές. Παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων και την κατάσταση στον τομέα της βιομηχανίας ένδυσης. Γνωρίζουμε ότι στις ε, ε, βιομηχανίες αυτές, ε, στον τομέα αυτό υπάρχουν συνθήκες οι οποίες καθόλου δεν συνάδουν με την σωστή κατάσταση και με που θα θέλαμε και όσον αφορά τους μισθούς και όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να στηριχτούν τα συνδικάτα και να υπάρξει διάλογος γόνιμος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει ε, την επίκλησή της ε, για ειρηνική επίλυση των διαφορών ε, μέσα από γόνιμο και επικοδομητικό διάλογο μεταξύ κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, καλωσορίζουμε την, το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των βουλευτών για το Λάος, έτσι όπως αυτό καταδεικνύεται μέσω του ψηφίσματος. κυρίως ε, όσον αφορά την ανεξήγητη εξαφάνιση του κυρίου Σόμπαθ Σόμχοουν ε, ήδη από τον ε, μήνα Δεκέμβριο του 12 αυτό εξακολουθεί να μας απασχολεί. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παρακολουθεί από κοντά το θέμα αυτό σε στενή επαφή με τις αρχές του Λάος. Το Λάος έδειξε κάποια διάθεση για διάλογο κύριε Πρόεδρε, αλλά δυστυχώς άνευ αποτελέσματος μέχρι τώρα. Όσον αφορά δε την διεθνή βοήθεια για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος αυτής της εξαφάνισης, μέχρι τώρα το Λάος έχει αρνηθεί. Σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και με τα κράτη-μέλη συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας. Ε, ευελπιστούμε ότι το Λάος ε, θα ε, προσυπογράψει την Διεθνή Συνθήκη για τους εξαφανιστέντες πρέπει να σας πω ότι ε, και με την χώρα αυτή έχουμε ε, διαρκή διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους κύριους δωρητές ε, του Λάος και έχουμε δει κάποια θετικά στοιχεία. Είμαστε βεβαίως πεπισμένοι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστώ κύριε Κάλλας. Έχουμε 7 ψηφίσματα για τη λήξη της συζήτησης και η ψηφοφορία θα γίνει μετά το τέλος της συζήτησης, στο τέλος του απογεύματος. Περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η κατάσταση για τις πρόσφατες εκλογές στο Μπαγκλατές. Η κυρία Κρόνπερ για 1,5 λεπτό μεταξύ των συντακτών της, ε, του θέματος, του ψηφίσματος. Ευχαριστώ. Πρόσφατα πάρα πολύ έχασαν τη ζωή τους έξω από την πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές